oh So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns fortfahren. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου επιτρέψετε να χαιρετήσω μία ομάδα επισκεπτών, 20 αν έχω ενημερωθεί σωστά, 20 ασκούμενοι της Γενικής Διεύθυνσης ε, σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Θα παρακολουθήσετε την ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν φαντάζομαι ότι είναι συνταρακτική για σας, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι ή μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσα η ψηφοφορία. Πάμε λοιπόν στην ε, εφαρμογή της, του Microfinance Facility. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Σούλτσε. Τροπολογία υπαριθμών 1, υπέρ παρακαλώ. Κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική α, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική β, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΒΑ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β' υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 12. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές Μισό λεπτό, καλύτερα να επαληθεύσουμε. Η 13 παρακαλώ, επαληθεύουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Αλλά ξαναψηφίζουμε μισό λεπτό για τη 13. Τροπολογία 13. Από ό,τι φαίνεται έχει χαλάσει η συσκευή του συναδέλφου μας. Ψηφίσατε όλοι. Αν δεν λειτουργεί η συσκευή του συναδέλφου, καλύτερα να καθίσει κάπου αλλού. και η Άγνες ε, θα κάτσει κάπου αλλού. Αν λειτουργούν όλες οι συσκευές, ας ξαναψηφίσουμε για την τροπολογία υπερθμών 13, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 16 υπέρ κατά ε, επανέλεγχος παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία απορρίφθηκε η 17 υπέρ κατά απορρίπτεται η 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η κοντ F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 21 υπέρ κατά επανέλεγχος Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοντ Α, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοντ Μπ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοντ Ε, υπέρ, κατά επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Η συμβαστική ή e υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην κοντ 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η κοντ 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η κοντ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 31 υπέρ κατά απορρίπτεται, η 32 υπέρ κατά απορρίπτεται, η 33 Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοντ 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοντ 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 35 υπέρ, κατά επανέλεγχος παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Η συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική σε α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η κοντ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 44 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 20 υπέρ κατά Νομίζω ότι ήταν η πλειοψηφία, ε, όμως παρόλα αυτά θα επανελέγξουμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική ή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην ε, τροπολογία 51. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 53 υπέρ κατά εγκρίνεται επαλήθευση για την 53 ψηφίσατε όλοι απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Και είστε συγγνώμη που δεν το είχα προσέξει. Η συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 58 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Η 60. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Η 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η κοντ 21. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Όχι, παρόλα αυτά, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 62 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Πάμε στην 64. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 67 παρακαλώ υπέρ κατά επαλήθευση παρακαλώ για την 67. Ψήφισατε όλοι, εγκρίνεται. 68. Υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά επανελέγχουμε την 68. Ε, Ψηφίσατε όλοι, εγκρίθηκε. Η 18, κοντ 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κοντ 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 71 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Η 72 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Η 73 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 75 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Η 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 77 υπέρ κατά εγκρίθηκε, η 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 79 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 79. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Οι 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 82 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε επαλήθευση για την 82 Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. 83 υπέρ. Κατά. Ε, και πάλι ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κοντ 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 85 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 86 υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Επαλήθευση 86 για την 86 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Αλλά το ΕΛΚ, στο ε, ΕΛΚ ψήφισε ένας παραπάνω. Μήπως μπορείτε να το δείτε λιγάκι. Απορρίφθηκε. Κόντεπτά, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 87 μισό λεπτό όχι αποσύρθηκε άρα η 88 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την 88 Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ε, κοιτάξτε, θέλω να με καταλαβαίνετε γιατί αυτή η αίθουσα ε, εδώ δεν βλέπει κανείς καλά και η άλλη αίθουσα είναι καλύτερη και γι' αυτό γίνεται συχνά επαλήθευση. Πάμε στην 89. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η κόντ 23, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η κόντ 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ μισό λεπτό μάλλον έχει καταπέσει 95 άρα πάμε στο 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 έχει αποσυρθεί άρα πάμε στην συμβαστική H στα αγγλικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η 99 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται η 25 κοντ 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κοντ 26 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται οπότε τώρα να ψηφίσουμε την έκθεση με ονομαστική βέβαια ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 49 υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Υποθέτω ότι δεν έχει κανείς αντίρρηση να προσθέσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην έκθεση. Ωραία, δεν βλέπω αντίρρηση. Θαυμάσια. Οπότε, οπότε, η επόμενη ψηφοφορία προς ε, μία πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Η συγγήτρια Γιούτα Στάινρουκ. Ε, είπε ο πρόεδρος Στάινμπρουκ που στα γερμανικά σημαίνει κάτι σαν πέτρινη γέφυρα αλλά λέει ότι δεν ήταν ένα κλασική φροηδική, ε, κλασικό φροηδικό λάθος. Συμβαστική F υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ υπέρ συμβαστική G παρακαλώ Ναι, λοιπόν, πρώτα θα ψηφίσουμε τη συμβαστική G. Πώς είπατε? Οπότε, οπότε. Λοιπόν, διαδικαστικά η γραμματεία μου διευκρινίζει ότι η προφορική τροπολογία είναι προσθήκη. Άρα πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβαστική G και μετά την ε, προφορική. Ο Σάνθος Κάζα έχει αντίρρηση. Τι λέει ο συγκεκριτής. Ο κύριος Κάζα. Όχι, πρώτα πρέπει να δούμε εάν η προφορική τροπολογία εγκρίνεται. Και αν εγκριθεί, τότε θα ψηφίσουμε τη συμβαστική μαζί με την προφορική τροπολόγησή της. Οπότε πρώτα πρέπει να δούμε τι είναι η προφορική τροπολογία, ποιος την προτείνει και μετά ψηφίζουμε την συμβαστική με την προσθήκη της προφορικής. Also gut, dann klären wir erstmal, ob es Widerspruch gegen das Oral Amendment. Λοιπόν, για να δούμε, υπάρχει αντίρρηση για την ε, προφορική τροπολογία. Α, υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχουν. Οπότε η προφορική τροπολογία απορρίπτεται, οπότε η διαδικασία είναι σαφής. Ψηφίζουμε τη συμβαστική G. Υπέρ παρακαλώ. Ωραία, κατά. Ωραία, εγκρίνεται. Οπότε, τροπολογία 24 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ έλεγχος για την 26 ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται Συμβαστική U υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά ας ελέγξουμε ελέγχουμε την 33 ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ Α, έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία για την J α. Α, βλέπω ότι οι σοσιαλιστές ε, είναι πανέτοιμοι. Ναι, φαίνονται να είναι 11 που χρειάζονται για να ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Ωραία. Οπότε κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική JA. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Λοιπόν, συμβαστική όμικρον. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Κ καπα λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ πρώτο τμήμα συγγνώμη πρώτο τμήμα της 105 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και είμαστε τώρα στην κάτι πρέπει να εξηγήσω. Ε, υπάρχει λάθος στο κατάλογο ψηφοφοριών. Για τη συμβαστική ΤΑΦ θα ε, προσθέταμε και την 124 που ε, εάν εγκριθεί η ΤΕ θα κατέπιπτε. Οπότε πρώτα να ψηφίσουμε την 125 υπέρ, κατά, αποχές και το τηλέφωνο σας παρακαλώ, ωραία. Λοιπόν, 125 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική ΤΑΦ. Οπότε ε, έτσι λίγο με και την 120 εγκρίνεται η ΤΑΦ, ωραία. Οπότε είμαστε συμβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε 144 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 147 σε τρία τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε 147 Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 26-26 απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα. 147 τρίτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Να ελέγξουμε και εδώ. Νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά... Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές. Ε, απορρίπτεται. 149 υπέρ. Α, καλά, να ελέγξουμε την 148. Επανερχόμεθα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Σαφέστατα. 149 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ζ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.

να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ με την προσθήκη μιας προφορικής ε, τροπολογίας. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη συμβαστική με την προσθήκη της προφορικής. ΑΒ με προφορική προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται 165 υπέρ Α είναι ταυτόσιμη την προηγούμενη ωραία συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 174 υπέρ κατά να ελέγξουμε 174 ψηφίσατε όλοι πέρασε ε συγγνώμη ε, απορρίπτεται τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 και 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συγγνώμη εγκρίνεται 180 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ψηφίσατε όλοι ευχαριστώ εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά απορρίπτεται. Περνάμε στην 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα ψηφίζουμε στην, για την το τελικό κείμενο άρχεται ψηφίσατε όλοι 48 υπέρ 4 κατά μηδέν αποχές συγχαρητήρια συγχαρητήρια στη συνάδελφου Στάιν Ρουκ δεν έχει κανείς αντίρρηση υποθέτω να προσθέσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο κείμενο ωραία όχι ωραία ωραία θα το προσθέσουμε Λοιπόν, να πω κάτι προσωπικό τώρα. Δεν θα έπρεπε να πω τώρα ότι ο Κέλερμαν μετά από 23 χρόνια συμμετείχε στην τελευταία ψηφοφορία του στην Επιτροπή μα. Δεν πρέπει να το πω, αλλά παρόλα αυτά το λέω. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο από πλευρά τη Επιτροπή μα. So, uh, Οπότε περνάμε στο σημείο 10 της μέρης διάταξης. Όιρες. Για το θέμα αυτό, ο έρθω Χάιντς Μπέκερ θα μας ε, παρουσιάσει συνοπτικά το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος γιατί θα πρέπει να κάνετε λίγη ησυχία, συνάδελφοι. Dominik. Okay, Heinz. vielen Dank, Herr Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να σας πω πού ακριβώς βρισκόμαστε. Σήμερα λοιπόν θα λάβει χώρα ο δεύτερος ε, τριμερής διάλογος και μεθαύριο ο επόμενος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μετά από συμφωνία με τους σκιώδης και με τη γραμματεία και με όλους ε, όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία με την νομική υπηρεσία και άλλους θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μέχρι τώρα ε, προχωρήσαμε ιδιαίτερα επικοδομητικά και μπορέσαμε να επιτύχουμε αρκετούς στόχους της Επιτροπής μας και αυτό μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ε, βέβαια δεν θέλω να προτρέξω γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια επίμαχα σημεία. Υπάρχει ας πούμε το θέμα του κατά πόσον θα συμπεριληφθούν οι κοινωνικοί εταίροι. Υπάρχει το θέμα των διασυνοριακών εταιρικών σχέσεων, των partnerships. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που εμάς μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Όπως σας είπα, μέχρι τώρα τα πάμε πολύ καλά, αλλά καλύτερα να το αφήσουμε να ολοκληρωθεί χωρίς να αγχωθούμε και μέχρι να ε, φτάσουμε και στις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις, που ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα ιδιαίτερα επίμαχο θέμα. περιπτώσει Επιτρέψτε μου με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδη ηγητές γιατί επικράτησε μεταξύ μας ε, ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία τους στόχους ε, τους, ε, επί των στόχων συμφωνήσαμε ομόφωνα και ελπίζουμε, ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπέκερ. Δεν ξέρω αν οι σκιώδη ηγητές θέλουν να λάβουν το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Άρα κακώς ανησύχησα που επικρατούσε ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, ο συνάδελφος Σάνων έχει το λόγο. Πολύ σύντομα. Να συμφωνήσω κι εγώ ότι η διαδικασία ήταν άκρος επικοδομητική, μεγάλη συνένεση και μέχρι τώρα τα πράγματα βαίνουν καλώς, άρα θεωρούμε ότι όσα έχουμε συμφωνήσει στην Επιτροπή μας ε, οι διάφορες πολιτικές ομάδες ότι θέλουμε να περιληφθούν στον λόγο νομοθέτημα. Μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο μέρος τους εμπεριέχονται στο νομοθέτημα και πηγαίνω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά για το Κοινοβούλιο. Αυτή ήταν δική μου σκέψη που ήθελα να την προσθέσω και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μπέκερ μιλάει στους τριμερείς διαλόγους τόσο καλά αγγλικά που ξέχασα σχεδόν ότι μιλάει γερμανικά. Φιλοφρονήσεις από ό,τι βλέπω, λέει ο πρόεδρο. Ηρωνικέ όμως εγώ θα τι χαρακτήριζα, λέει ο κύριο Μπέικερ. Ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μπέκερ και τους σκιώδεις και τους εύχομαι και στο μέλλον καλή συνεργασία. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 11. Ο κύριος Πυρίνσκι ζήτησε το σημείο αυτό να εξεταστεί ως το τελευταίο σημείο τη σημερινής διάταξη για να προσπαθήσει να είναι παρόν. Και όταν συζητούσαμε για τη μέση διάταξη, δεχτήκαμε αυτό του το αίτημα. Άρα δηλαδή πάμε στο σημείο υπαριθμών 12 απολογισμός της ε, τριμερούς κοινωνικής ε, συνόδου κορυφής. Η Άγνες Γιουγκέριος έχει παρακαλώ το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν η δεύτερη τριμερής κοινωνικής συνόδου κορυφής. Στείλαν παρατηρητή. Εγώ ήμουν συγκεκριμένα Είχαν τεθεί επιτάπτως πολλά ζητήματα, λίγο πολύ τα ίδια με όσα συζητήσαμε το πρωί με την Μαριάν Τάισεν. Βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης ε, του κοινωνικού διαλόγου, πώς ε, το REFIT και το καλύτερα νομοθετήν, το Better Regulation και ο κοινωνικός διάλογος ε, μπορούν να είναι επικοδομητικές διαδικασίες από κοινού. Συζητήθηκαν όλα αυτά. Συζητήθηκε πολύ επίσης και η συμβολή των κοινωνικών εταίρων σε ό,τι αφορά την υποδοχή των ετούντων άσυλο. και οι δύο πλευρές, ε, εργοδοσία και εργαζόμενοι, είπαν ότι αναζητούν τρόπους ε, για να βοηθήσουν στην ένταξη των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας. Υπήρξε επίσης ε, κάποια διαφορά από όσο και το περιεχόμενο της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα των εργαζομένων. Εκεί είδαμε να υπάρχει διάσταση απόψε μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Κάτι που θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα είναι ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ήταν παρόν, όπως και ο Ντόναλτ Τούσκ και δύο επίτροποι. Οι απερχόμενοι και η επόμενη προεδρία ήταν επίσης ε, εκπροσωπούμενες Το πώς οργανώνται όλα αυτά βέβαια ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα από πλευρά υλικοτεχνικής. Ε, επικράτησε κάποιο, κάποιο χάος. Πώς θα γίνει η κοινωνική ε, διάσκεψη κορυφής δύο ώρες. Προσπαθούν να οργανώσουν με διαφορετική σειρά από τη μία την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής και από την άλλη την σύνοδο κορυφής αυτή, αυτή καθεαυτή γιατί υπήρξε πρόβλημα με την οργάνωση. Ευχαριστώ. Έχετε παρατηρήσει σε από αυτού ίσως κάποιες ερωτήσεις να κάνετε από ό,τι βλέπω όχι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Κατόπιν τούτου πάμε στο επόμενο θέμα, σημείο υπερθμών 13 της ημέρης διάταξης, εφαρμογή της οδηγίας του συμβουλιου 2078 της 27 Δεμβρίου του 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Η συγγήτρια έρχεται, καθοδόν είναι. Γι' αυτό θα έλεγα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Λοιπόν, πέντε λεπτά διάλειμμα παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώ έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόβλημα. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Υπότιτλοι Jan Kunze. Jan. Jan Kunze. Jan. Παρακαλώ λες τους αδέλφους να γυρίσουν πίσω. setzen wir die Sitzung fort. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το σημείο υπαρχών 14 καλύτερα. Είναι οι πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό... Τα μπέρδεψα, λέει ο πρόεδρος. Προχώρησα μάλλον πιο κάτω από ό,τι έπρεπε. Όχι, ε, σωστά λέτε, έπρεπε να πάμε στο 13 και μέχρι τώρα απλώς ε, περιμέναμε την εισηγήτρια η οποία και ήρθε, η κυρία Ρενάτε Βίμπα. Και παρακαλώ έχετε και το λόγο κυρία Βίμπα. Κάνω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο εγγράφου εργασίας. που θα αποτελέσει τη βάση για το σχέδιο έκθεση το οποίο θα καταρτήσουμε στη συνέχεια. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το 2000 ε, οπότε και η εν λόγω οδηγία εγκρίθηκε ήταν ένα επίτευγμα, φανταστικό επίτευγμα θα το χαρακτήριζα τότε και είχε αναγνωριστεί ως επίτευγμα και από το, το πολιτικό κόσμο αλλά και από την κοινωνική, κοινωνία των πολιτών. 15 χρόνια μετά είναι ενδιαφέρον να δούμε πού βρισκόμαστε. Θέλουμε λοιπόν να αξιολογήσουμε την υλοποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 78 του 2000 για την ε, ισότητα στην απασχόληση καθώς επίσης και να υποβάλουμε συστάσεις. Όπως είπα, πρόκειται για το πρώτο σχέδιο του εγγράφου εργασίας το οποίο έχει την εξή διάρθρωση. Λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις που είχαμε από το 2000 και μετά. Η οδηγία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί από τα κράτη-μέλη τρία χρόνια μετά από την έγκρισή της. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πούμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. σε σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής. Πρόσφατα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, τα οποία δεν αφορούσαν συγκεκριμένα τις διακρίσεις, αλλά την αντίληψη που έχει ο κόσμος για τη διακριτική μεταχείριση. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν αποκαλύπτουν αύξηση διακριτικών συμπεριφορών και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός περισσότερο ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι υφίσταται διακριτική μεταχείριση ή τέλο πάντων παρατηρεί αυτά τα φαινόμενα. Η αύξηση ε, της διακριτικής μεταχείρισης πάντως φαίνεται να έχει αυξηθεί και δεν μιλάμε για τους τέσσερις μονολόγους που καλύπτονται εδώ, δηλαδή πεπιθήσεις, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, και σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτά τα τέσσερα καλύπτει οδηγία, αλλά υπάρχουν και για άλλου λόγου ε, συμπεριφορέ διακριτική μεταχείριση. Και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο από τι απαντήσει που έδωσαν οι ερωτηθέντε στο Ευρωβαρόμετρο. Δηλαδή, σε σχέση με την θρησκεία και τις πεπιθήσει, τα πιστεύω, υπάρχει αρκετά μεγάλη διακριτική μεταχείριση στα κράτη-μέλη. Όπως είπα λοιπόν, η διάρθρωση αυτό του εγγράφου εργασίας και αυτής της έκθεσης είναι η εξής. Πρώτον, θα εξετάσουμε το ζήτημα της έλλειψης ευαισθητοποίησης, συνειδητοποίησης και έλλειψης παροχής υποστήριξης στα θύματα. Τι θα πει αυτό, θα πει ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίο να γίνει δουλειά πάνω στην ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη για το τι εστί διακριτική μεταχείριση και τι δικαίωμα, τι δικαιώματα έχουν οι πολίτες. Δηλαδή ισότιμη μεταχείριση. Δεν ενώ συγκεκριμένα πολύ δαπανηρές αλλά ελάχιστα αποτελεσματικές ε, εκστρατείε πληροφόρηση, αλλά πιο πολύ συγκεκριμένε ενημερωτικέ εκστρατείε από στο μυαλό μου, οι οποίε θα μπορούσαν να δώσουν αυτά αποτελέσματα. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να παρέχεται υποστήριξη στα θύματα για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να πάψουν να νιώθουν θύματα. Να ξεπεράσουν αυτό το αίσθημα της θυματοποίησης. Επίσης, ό,τι αφορά ε, τα δεδομένα, την, ε, τα δεδομένα για την ποιότητα, για την ισότητα, συγγνώμη, ε, δεν απαιτείται συλλογή δεδομένων σε επίπεδο μελών και άρα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη διακριτικής μεταχείρισης αν δεν έχουμε στοιχεία για την ισότητα. Επίσης έχουμε χαμηλά επίπεδα καταγγελιών για περιστατικά διακρίσεων. Αυτό είναι το τρίτο κεφάλαιο της έκθεσης. Για αυτά τα χαμηλά επίπεδα υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πρώτα απ' όλα δεν αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι θύμα διατατική μεταχείρισης. Από την άλλη όμως, ένας άλλος λόγος είναι ότι υπάρχει ένα είδος νοοτροπίας, μια κουλτούρα, θα τη χαρακτήριζα, που λένε ότι και να κάνω καταγγελία δεν θα γίνει τίποτα, οι διαδικασίες είναι περιβολικά γραφειοκρατικές ε, και χρονοβόρες. Δεν υπάρχουν ε, και οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι. Με αυτά όλα θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και δύο ακόμη κεφάλαια που σχετίζονται μεταξύ τους. Το πρώτο είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Διότι σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι απαραίτητο να υπάρξει δίκη, ε, να υπάρξει προσφυγή στο δικαστήριο. Ένα ζήτημα λοιπόν που θα μας απασχολήσει είναι πώς οι εξειδικευμένες μη κυβερνικές οργανώσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν για τις ε, ορισμένες τουλάχιστον εκ των χωρών μελών βλέπουμε ότι όταν υποστηρίζονται τα θύματα από μη κυβερνητικέ οργανώσεις τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, είναι θετικά. Επίσης και για τα θύματα είναι πολύ ευκολότερο να συνομιλούν με άτομα από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σχετικό είναι και το κεφάλαιο παριθμών 5 που έχει να κάνει με τις κυρώσεις και τα μέσα νόμις προστασίας, τα ενδικά μέσα. Τα κράτη-μέλη έχουν εξειδικευμένους δημόσιους φορείς. Υπάρχουν δημόσιες αρχές, αλλά και αυτόνομα, ε, αυτόνομοι φορείς της ε, κυβέρνησης. Το θέμα είναι όμως η πρόσβαση σε αυτούς τους φορείς για αυτή την πρόσβαση πιστεύω ότι πολλά θύματα ε, χρειάζονται τη στήριξη από εξειδικευμένες με κυβερνητικές οργανώσεις. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι τι γίνεται σήμερα με την διερμηνία στα δικαστήρια. Πολύ σημαντικό είναι να βλέπουμε και τι ερμηνεία δίνεται από τα δικαστήρια και να την κοινοποιούμε γιατί είναι χρήσιμο για να αντιληφθεί ο κόσμος πώς τα δικαστήρια τα οποία επιλαμβάνουν των σχετικών υποθέσεων ερμηνεύουν τις σχετικές αυτές υποθέσεις. Και βέβαια το τελευταίο κεφάλαιο συστάσεις. Εν συντομία, αυτή είναι η μορφή που πιστεύω θα πρέπει να έχει έκθεση. Βέβαια, ευπρόσδεκτα τα σχόλια και υποδείξεις των συναδέλφων τις επόμενες εβδομάδες θα οργανώσω συναντήσεις με διάφορους φορείς, ΜΚΟ και άλλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, της καταπολέμησης δηλαδή των διακρίσεων, σε σχέση με την απασχόληση. Περιμένω τώρα να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Να δω τι έχουν να πούν για το θέμα. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Dann kommen... Πολύ ωραία. Ε, τώρα λοιπόν περνάμε στους ε, σκιοδησηγητές. Κυρία Ρατσέβιτς πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να συγχαρώ την ε, κυρία Βέμπερ, η οποία ξεκίνησε αυτή την έκθεση. Οι οδηγίες αυτές είναι 15 ετών, άρα είναι λίγο ξεπερασμένες. Όμως είχαν ε, μεγάλη σημασία για την αντίστοιχη νομοθεσία σε διάφορα κράτη-μέλη. Και οι δύο οδηγίες εφαρμόστηκαν μέσω κοινών κειμένων. Τα οποία βεβαίως έκτοτε έχουν τροποποιηθεί τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν πείρα από την εφαρμογή αυτών των νομοθετημάτων και έχουμε λοιπόν πολύ υλικό από την εφαρμογή αυτών των οδηγιών. Γιατί υπήρχε η απέτηση να υποβάλλονται εκθέσει για την εφαρμογή τη οδηγία κάθε μερικά χρόνια. Τακτικέ εκθέσει. Και γενικότερα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφοροι οργανισμοί που ασχολούνται με την ισότητα, μη κυβερνητικέ οργανώσει, η οργάνωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όλοι αυτοί έχουν εκπονήσει εκθέσεις. Έχουμε λοιπόν υλικό για την έκθεσή μας. Το έγγραφο εργασίας που λάβαμε είναι πολλά υποσχόμενο κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως ε, δεν περιγράφει απλώς τις οδηγίες, αναφέρεται στο ευρωβαρόμετρο, περιγράφει τη σημερινή συγκυρία και πλαίσιο. Όλοι παρατηρούμε αυτήν την ε, ενίσχυση των ε, ξενοφοβικών και ομοφοβικών τάσεων και ενεργειών που βεβαίως ε, σημαίνουν ότι αυξάνεται η ανάγκη να εξετάσουμε και να αντιμετωπίσουμε και πάλι το θέμα αυτό. Αυτές είναι λοιπόν οι πρώτες προτάσεις για να συμπληρώσουμε το ήδη υπάρχον και λειτουργικό πλαίσιο. Ούτω ώστε η εφαρμογή να γίνει πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πρακτικών, ε, εκπαιδεύσει των κεντρικών και περιφερειακών αρχών μελών, καθώ και κάλυψη των νομικών κενών αλλά και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έχουμε τεράστια πείρα από αυτά τα πράγματα. Διότι οι εκθέσει προόδου που έχουν εκπονηθεί ήδη έχουν αναφερθεί σε αυτές τις εκπαιδεύσει και στα κράτη-μέλη έχουν γίνει πολλέ εκπαιδεύσει και για του δικαστικού και για άλλου δημοσίου λειτουργού. Όλα αυτά είναι ουσιώδη για την σωστή ευαισθητοποίηση των αρχών για τις υποχρεώσεις τους περί ίσης μεταχείρισης. Φυσικά δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Η ευαισθητοποίηση βεβαίως πρέπει να είναι συνεχής. Πρέπει κατόπιν να ελέγχουμε ότι οι εκπαιδεύσεις αυτές ε, έχουν αποτελέσματα. Πιστεύω λοιπόν ότι η νομοθεσία μας θα πρέπει να ενθαρρύνει την οργάνωση τέτοιων εκπαιδεύσεων για να ε, γίνουν ευρύτερα γνωστές οι διατάξεις αυτών των οδηγιών. Χαίρομαι που ακούσαμε δηλώσεις ότι η έκθεση αυτή θα είναι αντικείμενο διαβουλεύσεων με διάφορους φορείς, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και εκπρόσωποι των εργοδοτών, διότι η έκθεση αυτή ε, τάσεται στεναρά στο πλευρό αυτών που μπορούν να υποστούν διακρίσεις, αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά την πλευρά των εργοδοτών που πρέπει να δημιουργήσουν το σωστό περιβάλλον για να μην υπάρχουν διακρίσεις στον τόπο εργασίας. Αυτό λείπει από την έκθεση. Και κάτι άλλο που λείπει στο κατάλογο αυτών των οποίων τη γνώμη πρέπει να ακούσουμε είναι κάθε είδους οργανώσεις των εργοδοτών. Το είπα ήδη. Τώρα για το περιεχόμενο της έκθεσης. Η δομή που προτείνεται είναι πολύ τεχνική και νομοθετική. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να τη συμπληρώσουμε με στοιχεία που ήδη αναφέρθηκαν και μεταξύ των νομοθετικών ε, θεμάτων που πρέπει να συζητήσουμε πολύ βασικό είναι να παρακολουθούμε την κατάσταση και να συλλέγουμε στοιχεία. Γιατί κάποια κράτη-μέλη τα συλλέγουν, αλλά όμως όχι. Στοιχεία για τις διακρίσεις. Και επίσης ε, η μετα-ανάλυση των στοιχείων μπορεί να γίνει μόνο αν τα στοιχεία αυτά είναι συγκρίσιμα. Άρα η συλλογή των στοιχείων και η πρωτοβουλία για αυτήν είναι πολύ σημαντική. Έχουμε λοιπόν 15 ετή πείρα και ξέρουμε ότι έχουμε τώρα νέες αντιλήψεις, νέα θέματα. Για παράδειγμα διακρίσεις μέσω διακρίσεων ε, εις βάρος οργανώσεων. Αυτά πρέπει να αναφερθούν πιο σαφώς. και ε, βεβαίως να καταγραφούν και στο νομικό τμήμα του κειμένου. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτό. Υπάρχουν και άλλες συστάσεις που είχαμε ήδη σε προηγούμενες εκθέσεις για να αυξήσουμε την, ε, αποτελεσματική, την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ε, των ε, φορέων που επιτηρούν την ισότητα στην πράξη. Και αυτά πρέπει να τα βάλουμε. Πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η Ρωμά έχουν αναφερθεί σε πολλές εκθέσεις ως μια συγκεκριμένη ομάδα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη συγκεκριμένα ούτως ώστε να μην υφίσταται διακρίσεις. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Βιτσιούτα. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο που μας παρουσίασε και θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει όλοι να συνεργαστούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την εφαρμογή της οδηγίας και να κάνουμε κάποιες ε, συστάσεις ε, που είναι απαραίτητο να τις προσέξουμε ιδιαίτερα. Έχουμε λοιπόν αξιολογήσει την έκθεση της Επιτροπής και εκθέσεις και άλλων θεσμών και βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα ε, στην εφαρμογή της οδηγίας. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να κάνουμε διαφορετική αξιολόγηση. Εγώ Πιστεύω ότι η συγγήτρια, η κυρία Ρενάτε Βίβα, έχει παρουσιάσει σωστά τη δομή της έκθεσης. Η δομή αυτή ε, μπορεί βέβαια να συμπληρωθεί αργότερα με το συγκεκριμένο περιεχόμενο της έκθεσης. Πάντως ε, θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο κατά πόσον τα κράτη-μέλη ε, καταθέτουν τις αληθινές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της έκθεσης. Γιατί δεν είναι προφανές, ε, δεν είναι σαφές ε, το κατά πόσον οι πληροφορίες είναι πραγματικές και δεν είναι εξοραϊσμός της κατάστασης. Μερικές φορές δεν είναι σαφές κατά πόσον μία περίπτωση είναι περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης ή όχι. Επίσης αυτό που μου αρέσει είναι η πρόταση της εισηγήτριας να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, ε, στα θύματα διακρίσεων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο θέμα αυτό και να καταθέσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Μία άλλη πρόταση που κατά την άποψή μου ε, μπορεί να είναι πιο σημαντική, δηλαδή ε, να καταθέσουμε κάποιες συστάσεις στα κράτη-μέλη, θεσμούς ε, και ΜΚΟ. Αυτό αφορά στην ανάγκη να διαδίδονται οι πληροφορίες και οι καλές ε, πρακτικές και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από εκείνα τα κράτη-μέλη όπου πράγματι υπάρχει εφαρμογή της οδηγίας και αυτές οι πληροφορίες θα τις ε, διαβιβάζουμε κατόπιν και στα υπόλοιπα, στα 28 κράτη-μέλη. Ε, εύχομαι λοιπόν ε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Χέλγα Στίβενς. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βέμπερ για τη θαυμάσια παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Καταλαβαίνω ότι στόχος της κυρίας Βέμπερ ήταν η υποβολή μιας πολύ αντικειμενικής πρότασης και συμφωνώ και με την άποψη του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη αυτά που έχει να μας πει και πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με το Φόρουμ για τις Αναπηρίες που είναι μια οργάνωση που από την αιγίδα της συγκεντρώνει πολλές οργανώσεις για τα άτομα με αναπηρία. Συνεργαζόμαστε με την Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Στηρίζω αυτά που ήδη περιέχονται στο κείμενο αλλά νομίζω ότι κάτι που είναι οσιώδες και που λείπει είναι να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα τις ανάγκες των ε, ατόμων με αναπηρία. Στο άρθρο 5 λέμε συγκεκριμένα ότι οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση και για τα άτομα αυτά. Τα μέτρα αυτά που διασφαλίζουν τη νοηματική διερμηνία και την αντίστοιχη κατάρτιση ούτως ώστε να μην υφίστανται τα άτομα με αναπηρία διακρίσεις. Ούτως άλλως ε, και η σχετική συνθήκη για τα άτομα με αναπηρία επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως λέει το άρθρο 5 για να αντιμετωπιστεί κάθε δυνατότητα διάκριση, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι θα γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές ε, στην νομοθεσία και πρακτική τους. Αυτό σημαίνει ότι και εδώ στην έκθεση πρέπει να αναφέρουμε το θέμα αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε μορφή διακρίσεων θα αντιμετωπιστεί για να μέγιστοποιήσουμε λοιπόν ε, το όφελος. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν οι ισχύοντες κανόνες πριν αναλυφθούν νέες πρωτοβουλίες. Προσβλέπω στη συνεργασία με την εισηγήτρια, στην περαιτέρω εργασία, για να διασφαλίσουμε ότι στα κράτη-μέλη και σε ενωσιακό επίπεδο θα σημειωθούν πρόοδοι για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ειρήνα Ρόνια Κάρη όμως δεν είναι εδώ. Η Τατιάνα Στάκοβα δεν είναι επίσης εδώ από τους Πρασίνους. Οπότε η Λάουρα Ατζέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την κυρία Βέμπερ για την εκθεσή της, για αυτά που μας είπε και όσον αφορά τα επτά σημεία τα οποία μας παρουσίασε. Θέλω να σας πω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε σύμφωνοι και όταν θα έχουμε το σχέδιο της έκθεσης ε, θα εκφραστούμε μέσω τροπολογιών και άλλων σκέψεων που θα θελήσουμε να καταθέσουμε. Εκεί ένα θέμα επί το οποίο συμφωνούμε ιδιαίτερα είναι ότι είναι απαραίτητο να ε, προβάλλουμε τα θύματα των διακρίσεων, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν υπήρξαν θύματα, να παρουσιάσουμε τα δικά τους τα δικαιώματα και το πώς είναι δυνατόν να στηρίξουμε τα θύματα αυτά στο να ζητήσουν αποζημίωση και γενικότερα αποκατάσταση. Αυτό είναι κάτι που μας βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνος. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ρόλο των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή είναι σημαντικό από την παιδική ηλικία να εξοικειώνονται τα παιδιά ευρέως και με δομημένο τρόπο για το ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων που μπορούν να καταστούν θύματα διακριτικής μεταχείρισης. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό να εξοικειωθούν τα παιδιά με όλες τις εκφάνσεις αυτού του φαινομένου. Εκτός από την οικογένεια υπάρχουν και άλλοι φορείς που νομίζω ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να προτείνω και άλλα δύο πράγματα που αφορούν στο πώς ακριβώς έχει αλλάξει η κοινωνία μας και κυρίως ε, του τι ισχύει σήμερα θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις ε, μεταναστευτικές ροές. Να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση όπου και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα θελήσουν να εργαστούν. Ε, θα πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να το λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας, γιατί πλέον η μετανάστευση και το μεταναστευτικό κίνημα αποτελεί εγγενές και αναπόσπαστο τμήμα των νέων γεωπολιτικών ε, καταστάσεων που επικρατούν στην Ευρώπη. Κάτι άλλο που θέλω να προτείνω και νομίζω επ' αυτόν θέλετε μπορούμε και να συζητήσουμε είναι το εξής. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ε, φυλακισμένους, τους έγκλειστους ε, σε φυλακές ε, στο χώρο εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί όταν αποφυλακιστούν, με ποιο τρόπο μπορούν να ενταχθούν στο χώρο εργασίας, πώς θα σου επιτρέψουμε να μπορούν και αυτοί να εργάζονται και μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι η φυλακή, η ποινή που τους επιβλήθη είχε ε, εκπαιδευτικό χαρακτήρα και κατόπιν μπορούν να ενταχθούν χωρίς πρόβλημα στο χώρο εργασίας. Ε, το λέω αυτό ε, κρίνοντας από τα δικά μας τα δεδομένα της Ιταλίας. Ξέρετε, αυτό στην Ιταλία δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα και γι' αυτό λοιπόν θέλω αυτό το θέμα να συζητηθεί. Επίσης ε, θα ήθελα να εκφράσω και τη δική μου εμπειρία να πω το τι ακριβώς κάνω εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω επερώτησης έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που όπως πολύ καλά γνωρίζετε καταδίκασε την Ιταλία γιατί δεν εφαρμόζει σωστά το άρθρο 5 της Οδηγίας 78 του 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί προβλέπεται για όλους τους εργοδότες ε, να ε, προσφέρουν ε, δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση στην εργασία, ακόμα και σε άτομα με αναπηρία. Άρα δηλαδή, παρότι έχουν περάσει, αν θέλετε, ε, σχεδόν 20 χρόνια, εντάξει όχι ακριβώς 20, 16 χρόνια, εξακολουθούμε ακόμα να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση έτσι ώστε να μην υπάρχουν ίσες συνθήκες πρόσβασης στην εργασία. Πολλοί δεν αναγνωρίζουν αυτό το δικαίωμα. Ε, άλλοι πάλι το θεωρούν δεδομένο. Αλλά ξέρετε, ένα δικαίωμα δεν πρέπει να την χάνει αναγνώριση. Ένα δικαίωμα πρέπει απλά να προσφέρει τη δυνατότητα να κάνει χρήση κανείς αυτού του δικαιώματος. Αυτό που με ενδιαφέρει το χάρη είναι εγώ να μπορώ να ασκώ αυτό το δικαίωμά μου, το να έχω πρόσβαση στην εργασία, το να το καταγγέλω, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Και μετά από 16 χρόνια, όπω σα είπα, η Ιταλία δεν εφαρμόζει το σχετικό άρθρο τη οδηγία. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με αυτά που λέει η κυρία Βέμπερ, ότι είναι απολύτω απαραίτητο να υπάρχει ένα διαρκέ feedback, μια αντίδραση από τα κράτη-μέλη σχετικά με την πρόοδο επ' αυτού του άρθρου. Ε, τελική ανάλυση τι νόημα έχει να ε, επεξεργαζόμαστε και να αποφασίζουμε επί κανονισμών τη στιγμή που αυτοί μετατρέπονται σε οδηγίες και αυτές κάπου χάνονται. Αυτό λοιπόν είναι εκείνο που μας ε, απασχολεί. Επ' αυτού θέλουμε να συνεργαστούμε, να συνεισφέρουμε κι εμείς και άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η Τατιάνα Στανόκα. Εντάξει, έχετε το λόγο, προηγουμένω δεν ήσασταν εδώ. Να συγχαρώ τη Ρενάτε για τις ε, προτάσεις της. Ε. Νομίζω ότι είναι καλή η δομή της έκθεσης όπως μας την προτείνει. Θα ήθελα ωστόσο να διτυπώσω κάποιες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά την έλλειψη που αναφέρατε, την έλλειψη δεδομένων. Ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Και εφόσον δεν διαθέτουν τα δεδομένα αυτά όλα τα κράτη-μέλη, αν τα διαθέτουν δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία με το σωστό τρόπο. Ξέρετε ότι κάποια κράτη τηρούν ε, υποχρεωτικά αρχεία, για παράδειγμα για την εθνική καταγωγή όπως στη δική μου χώρα τη Λετωνία. Άρα έχουμε διαθέσιμα στοιχεία και τα έχει αυτά τα στοιχεία η στατιστική μας υπηρεσία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για την ε, σύνταξη εκθέσεων και συλλέγει κάποια ε, στατιστικά στοιχεία επ' αυτών όλων. Έχω εργαστεί στο πλαίσιο της Επιτροπής πριν δύο χρόνια ε, για την τροποποίηση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τη συλλογή δεδομένων για την απασχόληση. Τα ad hoc modules συγκεκριμένα. Είχα προτείνει τότε λοιπόν δύο χρόνια πριν, είχα προτείνει στην Επιτροπή και στους κοιόδης εισηγητές να συμπεριληφθούν. Αλλά ως παρορετικά τα στοιχεία αυτά, στα ερωτηματολόγια. Λίγες όμως ήταν οι πολιτικές ομάδες που υποστήριξαν την ιδέα αυτή. Και δεν έγινε αποδεκτή στην ε, ψηφοφορία που είχαμε στην Επιτροπή. Αλλά κατ' εμέ αυτό είναι σφάλμα. Διότι αν θέλουμε να έχουμε δεδομένα, δεν είναι υποχρεωτικά βέβαια, αλλά και προαιρετικά να είναι. Αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει το πεδίο αυτό, για παράδειγμα, στο ένα ερωτηματολόγιο, σε ό,τι αφορά τι ε, τη ε, εθνική καταγωγή κτλ. Γιατί όχι, δεν θα έπρεπε να προβλέπουμε τη συλλογή στοιχείων. Δεν πέρασε τέλο πάντων αυτό, λυπούμε. Αλλά ελπίζω η έκθεση να τα καταφέρει καλύτερα. Θα την υποστήριξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ω τελευταία σκιώδη θα είχα δώσει το λόγο, στην κυρία Βιτσότου αλλά θα το δώσω στον Ντομινίκ Μαρτά που την ε, αντικαθιστά. Ευχαριστώ. Κυρία Βέμπερ, τι ωραίο θέμα. Η καταπολέμηση κατά των διακρίσεων. Αλλά για ποιες ε, διακρίσεις πρόκειται. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου κατά του πολιτικού ορθού και της ενιαίας σκέψης που έχει ως συνέπεια η καταπολέμηση των διακρίσεων να μετατρέπεται να γίνεται αυτό που τώρα αποκαλούμε θετικές διακρίσεις. Που τι σημαίνει στην πράξη. Προτίμηση για τους ξένους. Μέσω αυτής της καλλιέργειας της έννοιας, της μετάνοιας για τις ευρωπαϊκές χώρες που κάποτε είχαν ε, παγκόσμια σημασία καλλιεργούμε και το ξέρετε γιατί και εσείς στις χώρες σας και τις πόλεις σας και τις αγορές σας στις ε, ε, περιοχές στα προάστια που δεν υπάρχει δίκαιο Τι σημαίνουν όλα αυτά συγκεκριμένα για αυτούς που θέλετε να υπερασπιστείτε στην πράξη όλα αυτά μεταφράζονται σε διάθεση εκδίκησης. Εκδίκησης και στην πράξη πολλές φορές. Το βλέπουμε γραμμένο στους στίχους των εργατικών συνοικιών. Εντάξει, εντάξει, σας καταλαβαίνω, αλλά μην το παρακάνετε. Και φροντίστε παρακαλώ, φροντίστε να σκέφτεστε και τους συμπολίτες μας από τη δική μας εθνότητα που και αυτοί υφίστανται διακρίσεις και ρατσισμό. Προσέξτε κυρία Βέμπερ, προσέξτε. Και το ξέρετε. Με τέτοιου τύπου επιχειρήματα ο εθνικισμός, ο λαϊκισμός όπως τα αποκαλείτε, ξυπνάνε διότι τα μέλη της κυρίαρχης εθνότητας έχουν την εντύπωση ότι γίνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας την ίδια του τη χώρα. Λόγω αυτών των θετικών διακρίσεων που δίνει προτεραιότητα για την κατοικία, για την απασχόληση στις κοινωνικές παροχές, σε αυτούς που έρχονται από αλλού. Προσέξτε, προσέξτε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνάλφε, Μαρτά, μια προσωπική παρατήρηση. Επιτρέψτε μου. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε πόσα κύματα μετανάστευσης υπήρξαν στη Γαλλία τα τελευταία 100 χρόνια. Για τη Βαβαρία μπορώ να σας πω ότι τους τελευταίους αιώνες είχαμε 153 προσφυγικά κύματα. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να πει αν είναι ξένος ή ντόπιο. Δεν υπάρχει αυτή η διάκριση πιστεύω. Εγώ δεν ε, θεωρώ ότι είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας έναντι αυτών οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν πολέμους και έρχονται και ζητούν προστασία από μας. Αυτό ήταν μια προσωπική παρατήρηση. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης στις 25 Ιανουαρίου και στις 23 ε, Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και 16-17 Μαρτίου θα ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση εδώ ως Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο 14. Πολιτικές ε, ανάπτυξης δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή Μάρεκ Πλούρα. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Μάρικ Πλούρα. Παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να σας παρουσιάσω και εγώ το έργο μου για τις ε, πολιτικές ανάπτυξης δεξιτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Κατατέθηκαν μέχρι στιγμής περίπου 200 τροπολογίες και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες αυτές. Διότι οι τροπολογίες αυτές θα εμπλουτίσουν ε, την έκθεση. Να επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες ε, για κάποιους τομείς, αλλά να πω ότι υπάρχουν και κάποιες ε, ταυτόσιμες ε, τροπολογίες ή παρόμοιες τροπολογίες. Έχω ήδη ετοιμάσει 23 συμβιβαστικές τροπολογίες και τις έχω αποστείλει στους σκιώδεις εισηγητές και τους ε, συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Τον Οκτώβριο συνεδριάσαμε για να εξετάσουμε τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η συνεδρίαση διότι με τις συμβαστικές αυτές ε, τροπολογίες καλύπτονται πλέον 132, ε, τουλάχιστον από τις κατατεθείς τροπολογίες. Και καλύπτονται και όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Χάρη στη συμμετοχή των ε, σκιωδών εισηγητών νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου της έκθεσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τροπολογίες που καλύπτονται από τις συμβαστικές προτάσεις, ε, σε ό,τι περισσότερες τι περισσότερε, νομίζω ότι συμφωνούν με το πνεύμα της ε, έκθεση ε, και εμπλουτίζουν την έκθεση. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες τις οποίες δεν μπορώ να ρυθώ παρότι αντιλαμβάνομαι την πρόθεση των συντακτών τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τροπολογία του κυρίου Φουντούλη για τη μαθητεία. Ότι πρέπει να οδηγεί σε απασχόληση. Εγώ έλεγα ότι πρέπει, υπάρχει το should και το must. Ε, το must είναι πιο έντονη διατύπωση στα αγγλικά. Πρέπει να σας πω ότι συχνά ένας άνθρωπος ήταν πολύ νέος στην ηλικία και είναι ασκούμενος, εκπαιδεύεται, θέλει να αποκτήσει εμπειρίες, να κερδίσει και κάποια χρήματα. Αλλά η περίοδος μάθησης σε αυτή η άσκηση μπορεί να μην συμβαδίζει και εντελώς με την επαγγελματική σταδιοδρομία που θα ακολουθήσει στο μέλλον ο νέος αυτός. Γιατί πολλές φορές ε, την αξιοποιεί αυτή την περίοδο ένα νέο για να μάθει για τον εαυτό του, για ένα επάγγελμα και πολλές φορέ οι νέοι, ολοκληρώνοντα αυτή την περίοδο άσκηση, ή μαθητείας και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν θα τους ενδιέφερε να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες όπως η παριθμόν 91 ή η παριθμόν 52 για τις οποίες έχω κάποιες αμφιβολίες. Και αυτό όχι διότι διαφωνώ γιατί είναι εσφαλμένες ε, στο περιεχόμενό του απλά γιατί περιλαμβάνουν ε, υπερβολικές λεπτομέρειες και αφορούν τοπικά έργα, τοπικά project ή σε μη λίγες μόνο πηγές, συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Οπότε νομίζω ότι ουσιαστικά περιορίζεται έτσι ε, το πεδίο. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες όπως η περθμόν 64 και η 199 για παράδειγμα οι οποίες θεωρώ ότι παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας δεν συμφωνούν με τι αρμοδιότητε που έχουν τα κράτη-μέλη. Περί τροπολογία 59 τώρα, μπιτσότο. Ορισμό ευρωπαϊκών πολιτικών. Δεν με βρίσκει σύμφωνο ο ορισμό αυτό. Ούτε συμφωνώ ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι ένα lifting για να καλύψουμε το φιάσκο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ναι, μεν πιστεύω ότι πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν, ώστε οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ να βοηθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση της αγοράς εργασία σήμερα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για φιάσκο. Η αποκτήση δεξιοτήτων είναι πολύ ε, σημαντική. Ιδίω για την βελτίωση της κατάστασης ε, στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ και τώρα περιμένω να ακούσω τις απορίες σας. Ευχαριστώ. Vielen Dank. Jetzt wäre dran Petra Kumpula Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο θα είχε τώρα κανονικά η κυρία Πέτρα Νουπούλα, Νάτρη, αλλά δεν την βλέπω να είναι παρούσα. Κατ' ε, Κατά τούτου θα δώσω το λόγο στην κυρία Νάντια Τσιγκνάσκα από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Φλόρα για αυτή την έκθεση που μου φαίνεται πολύ καλή και χαίρομαι και για τη συνεργασία που υπήρξε για την εκπόνηση της. Να αναφερθώ σε τρία ζητήματα που θεωρώ σημαντικά. στο οποίο καταλήξαμε μετά από συμβασμούς, αλλά αναφέρονται και σε τροπολογίες που θα υποβληθούν για να βελτιώσουν, όπως είπε ο κ. Πλουρά, περαιτέρω το κείμενο. Πρώτον, σε όλα τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουμε ως φιλοδοξία η οι νέοι σε όλη, σε όλη τη ζωή να έχουν καινοτόμο πνεύμα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Όλοι θα πρέπει να επιθυμούμε και να στοχεύουμε να έχουν συγκεκριμένη πρακτική πληροφόρηση για το πώς να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, άρα να δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας. Όπως είπε και ο κύριος Πλούρα, η εκπαίδευση είναι βεβαίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε, βεβαίως να αναφερθούμε στο εκπαιδευτικό σύστημα και συμφωνώ ότι πρέπει να πούμε ότι όσοι έχουν πείρα από επιχειρήσεις αλλά και μη κυβερνικέ οργανώσεις αλλά και γενικότερα η κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχουν το λόγο τους για την εκπαίδευση. Αλλά πρέπει επίσης να επαϊπνούμε για να μην θίξουμε την επικουρικότητα. Κάτι άλλο που πρέπει να τονίσουμε. Δεν έχουμε επαρκέ προσωπικό, τουλάχιστον στη χώρα μου τη Σλοβακία. Δεν έχουμε αρκετού συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού. Το λέει και ο κύριο Πλούρα ε, στην έκθεσή του. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη βελτίωση τη ποιότητα του προσωπικού που βοηθάει. Ο κόσμος αλλάζει. Η αγορά εργασίας ε, αλλάζει επίσης με τρομερή ταχύτητα. Δεν έχουμε ιδέα πώς θα διαμορφωθεί σε μερικά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και τους ε, κατάλληλα καταρτισμένους και υψηλής ποιότητας ε, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Κάτι άλλο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η ομάδα των νέων με αναπηρία και των νέων που προέρχονται από μειονεκτικές ομάδες πληθυσμού. Πολλές φορές οι, οι δημόσιες πολιτικές δεν ασχολούνται με τους νέους αυτούς. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να έχουν και αυτοί κάθε δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους ε, γιατί μπορούν να κάνουν πολύ πιο δημιουργική την κοινωνία μας. Είναι πλούτος για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε περαιτέρω επ' αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα είναι παρούσα η κυρία Πέτρα Κομπούλα Νάτρη και παρακαλώ έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, θα μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι περισσότερο παρούσα εδώ, αλλά δυστυχώς η συνεδρίαση αυτή συμπίπτει και με άλλες, με την Ήτρε και λυπάμαι πολύ που δεν μπορούσα να είμαι ε, καθ' όλη τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια βάση ενόησης με τις ε, τροπολογίες μας, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε καλή έκθεση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης ε, όταν μιλάμε για την ανεργία των νέων. Και επίσης ε, πρέπει να πούμε ότι οι χώρες οι οποίες ε, αγωνίζονται με οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε δυσκολίες. Πολλές φορές αναγκάζονται να προβούν σε περικόπα στην παιδεία και ως εκ τούτου είναι πολύ πιο δύσκολο για τους νέου να βρουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είναι δύσκολο να βρουν δουλειά και αν δεν υπάρχουν πολλές θέσεις απασχόλησης, καταλαβαίνετε, αυτό πλήττει και τη νεολαία. Άρα δηλαδή η όλη αυτή η ιδέα πίσω από τα προγράμματα για τους νέους, πίσω από το πρόγραμμα Youth Guarantee είναι να βοηθήσουμε τους ε, ανθρώπους ε, που δεν έχουν δουλειά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Εγώ είμαι ανοιχτή για θέματα επιχειρηματικότητας, ε, και επίσης μπορούμε κάλλιστα να αναζητήσουμε και μια καλύτερη διατύπωση. Νομίζω ότι αν το καταφέρουμε αυτό θα αποτελεί επιτυχία για την Επιτροπή μας. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, ευπαθείς ε, ομάδες. Είναι σαφές ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Κάποιες ομάδες χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια. Η συνεργασία ανάμεσα στον στους εκπαιδευτικούς φορείς, τις εταιρείε και του ίδιους τους ε, νέους είναι καθοριστική σημασία. Εγώ διοργάνωσα ένα σεμινάριο επ' αυτού στη Φινλανδία ε, και τα πανεπιστήμια που ασχολούνται με εφαρμοζόμενες ε, επιστήμες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το πώς ακριβώς να χρησιμοποιήσουν τους ε, νέους επιστήμονες. Και αυτό είναι και μια πολύ καλή ιδέα και για να εκτιμήσουν και οι ίδιοι οι νέοι την ε, επιστήμη που σπούδασαν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιδέα. Βεβαίως ε, δυστυχώς δεν είναι εύκολο όλα αυτά, αλλά ως μητέρα κατανοώ ότι είναι πολύ σημαντικό ε, για, τα, για τους νέους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τους υπολογιστέ, τα τάμπλετ. Τώρα ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Η νέα γενιά είναι τελείως διαφορετική, πρέπει και αυτό να το δούμε. Και τέλος πιστεύω ότι και το εκπαιδευτικό σύστημα ε, θα πρέπει να καλύπτει όλους να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη νέα γενιά και για νέες δεξιότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος Ενρικε Σαμπόν, αλλά όπως το ξέρουμε ήδη, δεν μπορούσε να έρθει έτσι κι αλλιώς σήμερα το απόγευμα, ούτε και άλλοι συλλάδελφοι, η Λάμπερτ δεν είναι παρούσα, Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι και θα ήθελα να ευχαριστώ τη συνάδελφο ή μάλλον τον ε, εισηγητή για τη δουλειά που έγινε σε διάφορες συναντήσεις αναζητώντας συμβαστικές προτάσεις. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έλαβε υπόψη του τις δικές μας τις ε, προτάσεις και επίσης έλαβε υπόψη του και αυτά τα οποία ζητήσαμε που είναι σημαντικά θέματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η προσχολική εκκλησία η οποία, στην οποία έγιναν περικοπές είναι καθοριστική σημασία για την επιχειρηματικότητα. Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται από την παιδική ηλικία μέχρι την ηλικία που μπορούν να καταστούν επιχειρηματίες. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία σε βάθος ανάλυση και πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να αναζητηθούν μέθοδοι οι οποίες είναι αποτελεσματικές, να μην είναι όμως πιεστικές, ε, να μην ε, αγχώνουν τα παιδιά κατά την ανάπτυξή τους. Το θέμα της παιδείας είναι σημαντικό όπως σας είπα και για την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν κίνητρα στους νέους για να ακολουθήσουν αυτή τη σταδιοδρομία, τη σταδιοδρομία του επιχειρηματία. Υπάρχουν από την άλλη και τράπεζες που και αυτές μπορούν να παίξουν ρόλο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι οι μαθητείες, ε, τα τμήματα αυτά, ε, αυτές οι εκπαιδευτικές ε, μορφές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φτηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό είναι λάθος. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κατάλληλο εργαλείο γιατί όπως είπα και προηγουμένως η μαθητεία είναι καθοριστική σημασία για να ενταχθούν οι νέοι στον κόσμο της εργασίας. Βεβαίως ε, ε, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί δεν είναι δυνατόν να ξεκινάμε σήμερα ε, μια μαθητεία ένα τέτοιο σεμινάριο και στο τέλος ανακαλύπτω ότι δεν βρίσκω καμία θέση απασχόλησης. Πάντως, νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία να μην γίνεται κατάχρηση αυτού του εργαλείου, του εργαλείου της ε, μαθητείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και κάποια άλλα ε, που έχουμε σκεφτεί, ε, έχουν εκφραστεί, δεν εντάσσονται στους συμβασμούς, θα προσπαθήσουμε να τα αναφέρουμε. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσφέρουμε κάποιες εγγύσεις στους νέους, γιατί από τη στιγμή που βρίσκονται σε μία φάση όπου αναζητούν προσανατολισμό είναι πολύ σημαντικό να προστατεύει κανείς τους νέους, να τους προσφέρει εγγυήσεις για τις δυνατότητες που έχουν και για την κοινωνική προστασία την οποία μπορούν να απολαύουν τι είναι η δική μας η προσέγγιση. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει και κάποιος έλεγχος. Γιατί πολύ συχνά ε, ευκαιρίες που προσφέρονται από την Ευρώπη στα κράτη-μέλη, οι ευκαιρίες αυτές χάνονται, δεν προκύπτει αποτέλεσμα και αυτό γιατί δεν υπάρχει σωστός έλεγχος. Και αυτό είναι μια σημαντική προϋπόθεση. Και κάτι άλλο. Ε, είναι σημαντικό να ε, ελαφρυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φορολογικά ε, αυτό θα έχει άμεση σχέση με τους ε, νέους ε, άνεργους. Θεωρώ ότι κυρίως τα θέματα της φορολογίας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς κάποιες σκέψεις, κάποιο input για να αρχίσουν να γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρεται προηγουμένως ότι η τροπολογία που έχω καταθέσει για την δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ότι δηλαδή ε, πρέπει να καταβληθεί από τα κρατημέλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, ότι αυτό ε, είναι θέμα επικουρικότητας. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση όσον αφορά και δεν είναι δεσμευτική αυτή η τροπολογία. Εγώ θεωρώ όμως παρόλα αυτά ότι είναι θέμα πολιτισμού το να αποκλεί κανείς ανθρώπους από την παιδεία. Άρα δηλαδή θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν ε, σωστές προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι είπατε ότι είσαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε συζητήσεις για αναζήτηση συμβασμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ο Ντομινίκ Μαρτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συμφωνήσω σε όσους εξέφρασαν εγκόμιο προς τον κύριο Πλούρα στην Επιτροπή μας στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Νομίζω ότι είχα ήδη συγχάρει για το έργο του τον κύριο Πλούρα και μάλιστα τότε διακόπτει ο πρόεδρος. Με συγχωρείτε η γερμανική διερμηνία. Α, ωραία, ωραία. Τώρα έχουμε γερμανική διερμηνία. Συνεχίστε παρακαλώ. Να ξαναρχίσω από την αρχή. Ναι. Από όλα να τα ξαναπώ όλα. Λοιπόν, ε, συγχαρώ και εγώ τον κύριο Πλούρα για την εξαιρετική του δουλειά. Θυμάμαι και τα ξαναλέω, όπως είπα και πριν, ότι όταν μας παρουσίασε τον Ιούλιο την εκθεσή του συνεδρίασή μας ο κύριος Πλούρα, ήδη είχαμε εκφράσει την ικανοποίησή μας γιατί είχαμε πει ότι για όλους μας είναι προτεραιότητα η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Όμως, κύριε Πλουρά, είμαι απογοητευμένος τώρα, διότι ξέρετε καταθέσαμε πολλές τροπολογίες προς την σωστή κατεύθυνση, στο ίδιο πνεύμα με εσάς κύριε Πλουρά, θα περιστώ σε μία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν. Ουσιαστικά λέμε τα αυτονόητα. Δεν θυμίζουμε ότι πολλοί νέοι αναγκάζονται να δεχτούν επαναλαμβανόμενες περιόδους άσκησης που πολλές φορές αποτελούν συγκαλυμμένες μορφές ε, απα, ε, απασχόλησης ε, ή υποαπασχόλησης κατά κάποιο τρόπο. Δεν συμφωνούν όλοι οι παριστάμενοι με αυτή την τροπολογία. Νομίζω ότι τότε τον Ιούλιο το είχαν δεχθεί όλοι αυτό που είπαμε. Κύριε Πλούρα, γι' αυτό λοιπόν τώρα απογοητεύομαι. Ενώ υπήρχε συμφωνία, καμία από τι δικέ μα τροπολογίε δεν περιλαμβάνεται σε συμβιβαστικέ σα προτάσει. που σα προανέφερα ε, μία, η οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί συμβαστική τι, ταφ, αλλά δεν την έχετε συμπεριλάβει. Ξέρετε, εργαστήκαμε και μπορούμε και θέλουμε να εργαζόμαστε, αλλά ε, σε σχέση και με την προηγούμενη έκθεση, κύριε Πλούρα, ούτε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, παραλαμβάνω ότι τελικά βλέπω ότι εμεί είμαστε αυτοί οι οποίοι υφιστάμεθα πολιτική διάκριση εδώ. Δηλαδή, Όποτε ένας ε, βουλευτής από τη δική μας πολιτική ομάδα καταθέτει μια τροπολογία που λέει και τα ίδια με εσάς όμως τελικά κύριε Πλούρ. παρόλα αυτά απορρίπτεται αυτή η τροπολογία. Μόνο και μόνο επειδή προέρχεται από τη δική μας ομάδα, από το Front National. Εμείς λέμε τι ε, πιστεύουμε, συστηματικά όμως απορρίπτονται οι τροπολογίες μας, άρα υφιστάμεθα διάκριση και αυτό το θεωρούμε κρίμα. So, äh, ich nur Λοιπόν, τώρα και εγώ θεωρώ τις τροπολογίες που εγώ ο ίδιος κάνω είναι πολύ σωστές και ε, εκνευρίζομαι όταν δεν εγκρίνονται από άλλους. Δυστυχώς ε, η δημοκρατία είναι ε, το, το πολίτευμα όπου όλοι πρέπει να σέβονται την πλειοψηφία. Όχι, δεν θα το συζητήσουμε. Αυτή είναι η, προσωπική μου άποψη. Δεν θέλω να πούμε τίποτα περαιτέρω. Θα ψηφίσουμε για την έκθεση στις 3 Δεκεμβρίου. Οπότε έληξε και το 14. Φτάσαμε τώρα στο τέλος όπου έχουμε την έκθεση του κυρίου Πυρίνσκι για την αδήλωτη εργασία. Ο κύριος Πυρίνσκι όμως μπορεί να έρθει μόνο στις 6 και 4. δεν μπορώ να διακόψω για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τη συνεδρίαση. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν ότι στην προηγούμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο έγινε ένας τριμερής διάλογος που θα συνεχιστεί Η συνέχεια δεν δόθηκε τότε γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίε δικαιολογημένε. όμως δεν θέλω να σταματήσει η εξέταση αυτού του θέματος. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση από το θέμα αυτό και η Λουξεμβουργία στην Προεδρία. Θα ήθελε κατά τη διάρκεια της να έχει αυτή την έκθεση. Γι' αυτό θέσαμε το θέμα αυτό για σήμερα Όμως ε, θα το βάλουμε στις 27 Νοεμβρίου, 9.30 με 12, τότε θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Και ελπίζουμε τότε να σας παρουσιάσουμε και κάπως αναλυτικά και τις τρεις αποστολές Πορτογαλία, Ολλανδία και Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σήμερα, επειδή είχαμε τη συζήτηση με τη Μαριάννε Τάισεν, αναβάλαμε το θέμα αυτό. Η επόμενη συνεδρίαση, λοιπόν, σημειώστε παρακαλώ προσωρινά έκτακτη συνεδρίαση στις 27 Ενδεκάτου 9.30 με 12 και η επόμενη τακτική συνεδρίαση θα είναι στις 3 Δεκεμβρίου 9 με 12.30 και 2 με 5.30 εδώ στις Βρυξέλλες οπότε εξαντλήσαμε την σε διάταξη σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας ευχαριστώ και του διερμηνείς Δεν νομίζω πως θα συνοχωρηθούν που κλείνουμε νωρίτερα τη συνεδρίαση. Έχω μια μισή ώρα για να ασχοληθούν με άλλα εποφελή θέματα. Καλό σας βράδυ.